Στην δεκαετία του 80 κύριε Επίτροπε όταν εσείς επισκεπτόσασταν το Τσερνομπίλ είχε συνταχθεί ένας νόμος με μία ρήτρα αναθεώρησης. Πότε λοιπόν θα έρθει αυτή η αναθεώρηση? Σας ευχαριστώ κύριε Μπελέτ. Ε, ολοκληρώνει την εξέλιξη του θέματος αυτού. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο το μεσημέρι στις 12. Το επόμενο θέμα της τη έρεξη είναι η δήλωση της Εκτελεστικής Επιτροπής για πρακτικές πτυχές αναθεώρηση των μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδοτική στήριξη των ΜΜΕ κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Το λόγο θα, θα έχει ο Επίτροπος Ταγιάννη πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με ποιο τρόπο η Κομισιόν προτίθεται να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να, αυτοχρηματο... να χρηματοδοτηθούν ούτως ώστε να μεγαλώσουν. Εμείς στα πλαίσια του 2020 υποσχεθήκαμε να βασιστούμε στην ανάπτυξη που θα βασίζεται στη γνώση και στην κοινοτομία. Οι επιχειρηματίες που ξεκινούν νέες επιχειρήσεις, ε, δημιουργούν νέες ε, ιδέες, δημιουργούν και νέες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Εμείς θα πρέπει να προσπαθήσουμε αυτές οι επιχειρήσεις να έχουν και τους απαραίτητους πόρους και τη χρηματοδότηση πιο συγκεκριμένα για την κοινοτομία. Διότι θα συνεχίσω να το επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν υπάρχει ανταγωνιστικότητα, δεν υπάρχει κοινοτομία. Πρώτα απ' όλα, εμείς τις προτάσεις μας ε, θέλουμε να υπογραμμίσουμε την σημασία της έρευνας και της καινοτομίας. Όπως αναφέρεται στην πράσινη βίβλο της ε, Κομισιόν που εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας, θέλουμε να απλωστεύσουμε την λειτουργή, τη διαχείριση αυτών των προγραμμάτων μέσα από τη διαχείριση κοινών σχεδίων σε συνεργασία με τους εταίρους μας και θα εγγυηθούμε έτσι και μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά. Απλούστευση και ευελιξία λοιπόν. Θα είναι δύο λέξεις κλειδί των μελλοντικών μας εργασιών. Που στοχεύουν στην πρόθεση της ανάπτυξης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα προγράμματα και τα κοινοτικά μέσα θα πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και σε όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που έχουν προπτικές ανάπτυξης. Οι ΜΜΕ θα πρέπει να συσπηρωθούν μέσα σε ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα καταγράφει όλη την κεκτημένη εμπειρία. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις αλλαγές των αγορών κατά την επόμενη περίοδο δημοσιονομικού προγραμματισμού. Επίσης πρέπει να δούμε ποια θα είναι τα χρηματοπιστωτικά μέσα από την επιδότηση στα δάνεια προς τις επιχειρήσεις. Αυτό φυσικά για όποιον θα μας έρθει με ένα επιχειρησιακό σχέδιο, ένα business plan λογικό. Να δώσουμε εγγύσεις και επενδύσεις με κεφάλαια κινδύνου. Αυτά τα μέσα μας βοήθησαν να πετύχουμε πολλά πράγματα. 100.000 επιχειρήσεις μέσα από αυτό το πρόγραμμα βοηθήθηκαν και όταν θα θα φτάσουμε στο τέλος του προγράμματος, θα έχουμε βοηθήσει πάνω στις 300.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. και το 98% του επενδεδημένου κεφαλαίου δεν έχει ακόμα επενδυθεί. Με μόνο με το 2% βοηθήσαμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Και δεν πρόκειται εδώ για γραφειοκρατικά μέσα. Πρόκειται για κονδύλια τα οποία τα παίρνει κανείς στην τράπεζα. Δεν μπορεί δηλαδή να Δεν, δεν χρειάζεται να έρθει να τα ζητήσει στις Βρυξέλλες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εκτιμούν ιδιαίτερα την αποτελεσματικότητα αυτών των σχεδίων. Πριν από λίγες μέρες το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από την Κομισιόν να δημιουργήσει ένα καθεστώς κεφαλαίων κινδύνου σε κοινοτικό επίπεδο. Ερχόμαστε λοιπόν να καλύψουμε το κενό των αγορών. Επίσης, Έχουμε και το καθεστώς εγγύησης των δανείων που βοηθά ιδιαίτερα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Κομισιόν είναι πεπισμένη ότι οι εγγύησει για τα δάνεια είναι απαραίτητα και σε περιφερειακό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα δημιουργήσουμε λοιπόν εμείς όλα αυτά τα μέσα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καλούμε... Καλούμε λοιπόν όλα τα κράτη τα οποία συναποφασίζουν μαζί με μας για αυτά τα θέματα να μας βοηθήσουν για τη μελλοντική δημοσιονομική φάση. Πρέπει να προσθέσω ότι στο μεταξύ η Κομισιόν δεν έμεινε με δεμένα χέρια. Στις 28 Σεπτεμβρίου συναντηθήκαμε με το στο φόρουμ το ΜΜΕ για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τις καλύτερες πρακτικές και να μπορέσουμε να ενθαρρύνουμε νέες λύσεις. Αυτό το μόνιμο φόρουμ συσπηρώνει τακτικότατα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση της αγοράς και το νομικό πλαίσιο για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Συζητιούνται επίσης και διάφορες εφαρμοστικές λεπτομέρειες και προχωράμε ιδιαίτερα. Εξίσου σημαντικό είναι να δούμε ποιο είναι και το ρυθμιστικό πλαίσιο. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον συνάδελφο Μισελ Μπαρνιέ που προτείνει πολλές πρωτοβουλίες που καθιστούν ιδιαίτερα αποτελεσματικές τις, νομοθε... τις δικές μας νομοθεσίες και το δικό μας σχεδιασμό κυρίως για τα κεφάλαια κινδύνου, για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματικότητα. Τώρα, για τα περιουσιακά στοιχεία των ε, τραπεζών Βασιλεία 3. Η Κομισιόν θα εκπονήσει το Ιούλιο του 2011 τις νομοθετικές προτάσεις. Θα έχουμε μία αξιολόγηση των μικροοικονομικών και μακροοικονομικών επιπτώσεων αυτών των διατάξεων. Και θα θέλαμε λοιπόν οι προτάσεις σας να είναι ιδιαίτερα εύστοχες λαμβάνοντας υπόψη τι γίνεται και αλλού ανά τον κόσμο. Για να ολοκληρώνω, πρέπει να πω ότι οι δημαρχές του προϋπολογισμού θα είναι αυτές που θα αποφασίσουν για όλα αυτά τα μέτρα και τον προγραμματισμό. Σε αυτή τη φάση η λιτότητα είναι όσο το δυνατό, χρειάζεται όσο το δυνατόν καλύτερα να ξοδευτούν αυτά τα χρήματα. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε κίνητρα και για την ιδιωτική χρηματοδότηση. Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ούτω ώστε οι προτάσεις μας να επικεντρώνονται ιδιαίτερα στη σημασία της ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για το μέλλον της Ευρώπης. Πεπισμένοι όπως είμαστε δηλαδή ότι όλη, οι όλη η δουλειά που πρέπει να κάνουμε στο μέλλον για την ανάκαμψη της μεγάλης βιομηχανίας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της και την ανάπτυξη των ΜΜΕ που είναι αυτές που μπορούν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και τις κοινωνικές πτυχές και να, και συνεισφέρουν στην επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στον κοινωνικό τομέα. Για να μπορέσουμε να λιάνουμε το έδαφος και να ξεκινήσουμε την επόμενη φάση μετά την κρίση. Ευχαριστώ κύριε Ταγιάννη. Τώρα θα ακούσουμε τους ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Πρώτος ο κύριος Μπέντσεν εξ ονόματος του ΕΛΚΑ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Ταγιάννη για όσα μας είπε. Το θέμα αυτό το θέσαμε σήμερα στην ημερησία διάταξη γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σημαντικότερο από ποτέ να εξετάσουμε το θέμα της χρηματοδότησης των ΜΜΕ στην Ευρώπη δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι ΜΜΕ έχουν περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και ότι αυτό είναι εμπόδιο για την ανάπτυξη αυτών των επιχειρήσεων και για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Και αυτό βέβαια διαφάνει ακόμα πιο ξεκάθαρα μέσα στα πλαίσια της ε, χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότηση από τις τράπεζες στην Ευρώπη η εξάρτηση από τις τράπεζες στην Ευρώπη είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στην Αμερική και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει διακανονισμός βάσει της Βασιλείας 3. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι θα υπάρξουν ακόμα μεγαλύτερες ε, δυσκολίες όσον αφορά τη συμμετοχή στον κίνδυνο των ΜΜΕ όταν έχουμε τη Βασιλεία 3. γιατί το κεφάλαιο που διατίθεται από τις τράπεζες σημαίνει ότι είναι πολύ ακριβό. Και αυτό σημαίνει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν προβλήματα και υπάρχει απώλεια θέσεων απασχόλησης. Θα πρέπει να ενδυναμώσουμε εκείνα τα μέσα που συμβάλλουν στην ε, ανάπτυξη και την καινοτομία των ΜΜΕ. Και θα ήθελα ακριβώς να σας πω ότι θα ήταν καλό να ε, εμπλακούμε πολύ περισσότερο για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις ΜΜΕ. Τα προγράμματα αυτά αφορούν την πρωτοβουλία της, ε, που θα μπορέσει να βοηθήσει τις ε, ΜΜΕ. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα, ακόμα και το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο μπορεί να βοηθήσει εδώ και γι' αυτό είναι σημαντικό να πούμε ότι θα πρέπει να συγκεντρώσει την προσοχή του το Κοινοβούλιο του επόμενου μήνε σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Θα ακούσουμε την κυρία Χέρτσοβ, εξονόμητο των συσχελιστών τώρα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε Επιτροπέ, θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα κι εγώ σήμερα ούτω ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσει στην πατρίδα μου τη συζήτηση. Όταν ε, γινόταν η συζήτηση των τριών στόχων του πακέτου, τι ακούσαμε, ότι το ε, ότι θέλουμε να ε, εισέλθουν στην αγορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως με νέα προϊόντα. Δεύτερος στόχος, μείωση της γραφειοκρατίας και εξαιρετικό παράδειγμα βέβαια είναι και η σχετική οδηγία για τις υπηρεσίες. Τρίτον, Τρίτος στόχος ήταν ε, η διευκόλυνση της, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως προς τη χρηματοδότηση, να βρούμε νέα μέσα χρηματοδότησης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παράγουν το 1 τρίτο του ΑΕΠ. Ε, Εάν λοιπόν εξετάσουμε το θέμα από αυτή την πλευρά, διαπιστώνουμε ότι συμβάλλουν κατά το 1 τρίτο στον προπολογισμό ε, τη Ένωση. Α δούμε όμω το τμήμα του ε, προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση που αφιερώνει τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Σίγουρα δεν μπορούμε να δηλώσουμε ικανοποιημένοι με την αναλογία. Ε, τραπεζικά είχε και έχουν λάβει εκατοντάδε επιχειρήσει ε, πέρυσι, ε, αλλά δοθεί εκατοστέντος ε, του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 23 εκατομμύρια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι είναι ε, αυτές οι εκατοντάδες ε, οι 100.000 ζητώ συγγνώμη εγγυήσεις που εδόθησαν. Εντάξει, θα μου απαντήσετε ότι πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις είναι, εμπλέκονται σε δραστηριότητες υψηλού κινδύνου, venture capital, αλλά αυτό δεν είναι πλήρη απάντηση. Χρειαζόμαστε, Επίτροπε, ένα πακέτο το οποίο ε, θα καθιστά δυνατή την ε, ευέλικτη και αποτελεσματική χρήση των χρηματοδοτικών μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας ε, για την και πρέπει να καλέσουμε τα κράτη-μέλη να αναλάβουν δράση και όχι να μένουν στα λόγια λέγοντας ότι υποστηρίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σας έχουμε στείλει μία επιστολή για αυτό το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σας παρακαλώ, σας το λέω και τώρα, μην ξεχνάτε Αυτέ τις επιχειρήσεις γιατί είναι στη δυσχερέστερη θέση μετά από τα μέτρα λιτότητα που υιοθέτησαν ε, τα κράτη-μέλη. Ταυτόχρονα όμω, αυτές είναι επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις απασχόληση. Το Κοινοβούλιο οφείλει να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο κύριος Σμί τώρα από πλευρά των ε, Φιλελευθέρων και Δημοκρατών. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε, καλά κάνουν, κάνει η Επιτροπή και είναι φιλόδοξη, ε, διότι είναι σαφές ότι είναι πελώρια η πρόκληση στην οποία καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε. Έχουμε 20 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αντιστοιχούν στο 99% του συνόλου των επιχειρήσεων ε, και ε, λέει ο Επίτροπος ότι είναι ο γίγαντας ευρωπαϊκής οικονομίας οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτό αληθεύει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να μεγαλώσουν αυτές οι μικρομεσαίε επιχειρήσεις. Πώς θα μεγαλώσουν, χρειάζεται χρηματοδότηση, όπως είπαν και οι συνάδελφοι. Όπως είπε και ο Επίτροπος, με τα νέα μέσα χρηματοδότησης, δηλαδή να δημιουργήσουμε τι υφιστάμενε δυνατότητες χρηματοδότησης και να ε, χρησιμοποιήσουμε παραδείγματο χάρη τα διαρθρωτικά ταμεία και τα κονδύλια που υπάρχουν εκεί. Όπω είπε και ο κύριος Μπένσεν νωρίτερα, οι ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, έχουν πάρα πολλά συμφέροντα μέσα σε αυτόν τον κανονισμό. Εδώ έχουμε φτιάξει χιλιάδες κανόνες για το χρηματοπιστωτικό τομέα. Οι περισσότεροι χρειάζονται. Αλλά σίγουρα με αυτούς τους κανόνες αυξήθηκε το κόστος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να μπορέσουν να συνάψουν δάνειο. Ε, και ε, σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουμε επίγνωση ακριβώς ποιος είναι ο τελικός λογαριασμός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σα παραπέμπω και στι απαιτήσει ε, τη ε, Βασιλεία 2 ε, για τι επιχειρήσει αυτέ. Χρειαζόμαστε ευελιξία για τα μέσα χρηματοδότηση και πρέπει αυτό να είναι το βασικό στοιχείο, να καταργήσουμε την γραφειοκρατία. Επίτροπε, μπορείτε να βάλετε το χέρι στην καρδιά και να μα πείτε ότι ειλικρινά πιστεύετε πω αυτή είναι η λύση για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, Δηλαδή πιστεύουν, πιστεύει το προσωπικό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ότι αυτό κάνει η Ένωση, ότι βελτιώνει την κατάσταση ή το αντίθετο να αυξάνει τη γραφειοκρατία. 20 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις είπαμε έχουμε στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και 20 εκατομμύρια ανέργους ε, στην Ευρώπη. Και αυξάνεται ο αριθμός, αυξάνεται η ανέχεια, αυξάνεται η φτώχεια για να τα καταφέρουμε. Εμείς, και όταν λέω εμείς, όλοι εμείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινηθεί ούτω ώστε με πυγμή να προωθήσει αυτά τα νέα μέσα χρηματοδότηση, να στηρίξουμε αυτέ τι επιχειρήσει, γιατί εκεί φτιάχνονται οι θέσει εργασία τη Ευρώπη. Σα ευχαριστώ. Ε, από του συντηρητικού και μεταρρυθμιστέ, ο κύριο ε, Τσβαρνέσκι, παρακαλώ. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, συζητάμε για ένα τομέα τη ε, οικονομία που έχει βασική σημασία. Πρόκειται μια ΜΜΕ, οι οποίες είναι εκείνες που ε, δίνουν τις περισσότερες θέσεις απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο σύνολο. Πολύ περισσότερες από ότι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Είναι μικρές οι επιχειρήσεις αυτές πολλές φορές είναι οικογενειακές και επλήγησαν περισσότερο από τις επιπτώσεις της ε, οικονομικής κρίσης. Ακόμη περισσότερο, ε, το ε, κοινωνικό κόστος της αποδυνάμωσης του τομέα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, οι μεγάλες εταιρείες και τα μεγάλα βιομηχανικά λόμπι είναι πιο αποτελεσματικά στην προάσπιση των συμφερόντων τους αλλά θα πρέπει να προασπίσουμε και τις ΜΜΕ γιατί αυτό σημαίνει ότι θα προασπίσουμε τους φορολογούμενους και τους πολίτες των κρατών μελών. Και δύο λόγια ακόμα. Θα ήθελα να τονίσω ότι τα κράτη-μέλη δεν πρέπει να κατηγορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση για οτιδήποτε. Θα πρέπει να ασχοληθούν με το να προσπαθεύσουν τις ΜΜΕ και συμφωνώ με αυτά που είπε η κυρία Ευχαριστώ. Ο κύριος Μορκάντη. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, τα τελευταία χρόνια και έγινε, γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσουν να παίρνουν δάνεια και αυτό και λόγω της ε, κρίσης. Στον προγραμματισμό της ε, Κομισιόν βλέπουμε να έχουμε σημαντικά κενά βλέπουμε να υπάρχει μια διάχυση στις γραμμές παρέμβασης. Με το νέο προγραμματισμό για τις ΜΜΕ θα πρέπει να απλουστεύσουμε τους κανόνες που δυσκολεύουν κυρίως τις μικρές επιχειρήσεις. Θα πρέπει να έχουμε δε μια ενιαία θηρίδα για την πρόσβαση στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Θα πρέπει να έχουμε νέα μέσα νέα οικονομικά μέσα που θα βοηθούν την πρόσβαση στις, στα δάνεια, που θα ευνοούν την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει να διευκολύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την ζωή αυτή της πραγματικότητας ε, στην Ευρώπη που απασχολεί πάνω από 300 εκατομμύρια άτομα και που είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο κύριος Στογιάνοφ για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Όπως και προλέσσαντες, θα ήθελα κι εγώ να πω ότι συμφωνώ με αυτά που είπανε για τις ΜΜΕ. Συμφωνώ αυτό που είπαν οι συνάδελφοι μέχρι τώρα, ότι δηλαδή οι ΜΜΕ είναι εκείνες που υπέφεραν περισσότερο από την οικονομική κρίση. Και το είπε και ο κ. Σονέτσκι αυτό με τον οποίο μπορώ να συμφωνήσω πολλές φορές είναι οι οικογενειακές επιχειρήσεις αυτές πάρα πολύ μικρές οι οποίες όμως βοηθούν στην επιβίωση μιας οικογένειας. Λοιπόν, εμείς βοηθάμε μια μεγάλη επιχείρηση που πλήττεται από την ε, οικονομική ε, κρίση και η οποία έτσι καταφέρνει να έχει κέρδος. Όταν όμως πληγεί μία μία έψιλον, ε, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τα προστοζήν. Οι μεγάλες επιχειρήσεις πλήττονται μόνο αν πληγούν στο κέρδος τους. Θα πρέπει λοιπόν να πω ότι ορισμένες τροπολογίες που υπευλήθησαν μπορεί να έχουν ανητικέ επιπτώσεις. Δηλαδή οι τραπεζικές εγγύσεις δεν θα ήταν επαρκές. Πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν περισσότερος διακανονισμός βέβαια του τραπεζικού τομέα και θα πρέπει να μπορούν έτσι να δοθούν περισσότερα κονδύλια στις ΜΜΕ γιατί πιστεύω ότι δεν μπορούμε να θέσουμε επίσης όρες τις μικρές και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν οι μικρέ επιχειρήσει να είναι για εκείνε ανταγωνιστικέ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Ένα άλλο λεπτό, κύριο Ρίμπεκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Επίτροπε, καταρχήν θα ήθελα να σα ευχαριστήσω. Γιατί ακριβώς το πρόγραμμα ΣΥΠ αυτή τη στιγμή είναι ένας πυλώνας. Το ίδιο ισχύει και για τα προγράμματα Ζερεμί, Ζασμίν, και εράσμους για νέους επιχειρηματίες γιατί αυτό συμβάλλει στην ε, γνωριμία των αγορών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Χερτσόκ που αναφέρθηκε στο στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Αυτό που θα ήθελα να εκφράσω όμως είναι μια παράκληση προς τον Επίτροπο Ταγιάννη. Στους στόχους ε, για το 2020 θα πρέπει να φροντίσουμε οι ΜΜΕ να έχουν μια ελάχιστη κεφαλική κάλυψη της τάξης του 20% όπως ζητάμε από τις τράπεζες το ίδιο πρέπει να κάνουμε και από τις ΜΜΕ και επίσης θα ήθελα να πω ότι ε, η φορολόγηση του κέρδους θα πρέπει να γίνεται μόνο εάν τα χρήματα αυτά αποσύρονται από την επιχείρηση Εάν χρησιμοποιούνται για την ενδυνάμωση επιχείρηση δεν πρέπει να φορολογούνται. Και τελευταίο σημείο που είναι σημαντικό, η δυνατότητα έκπτωσης από τους φορούς δεν θα πρέπει να είναι κάτω από τις 5.000 ευρώ. Αυτή ήταν η καλύτερη βάση νομίζω, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε ίδια κεφάλαια και κεφάλαιο κινδύνου για την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αυτών. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Ρουμπίκο. Ο κύριος Κούτας έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα πρέπει να σκεφτούμε και να βασιστούμε στις ευρωπαϊκές αρχές. Το 2 τρίτο των θέσεων σχόλες στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργούνται από τις ΜΜΕ. Υπό τους όρους της ε, τωρινής κρίσης η πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση είναι όμως πάρα πολύ δύσκολη. Δεν είναι ιδιαίτερα γενναιόδρες οι τράπεζες. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την πρόσβαση στην ε, χρηματοδότηση και στην ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Υπάρχουν δυσκολίες όσον αφορά την ενημέρωση της πρόσβασης ε, στα Ταμεία Επενδύσεων και έλλειψη διοικητικών ε, δυνατοτήτων για να μπορούν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες αυτές. Ε, μεταξύ των ετών 2014 και 2020 θα πρέπει να δημιουργηθεί καλύτερη διαφάνεια μεταξύ τραπεζών και επιχειρήσεων, καλύτερη ενημέρωση όσον αφορά τις δυνατότητες που υπάρχουν και τις δυνατότητες ε, δανειοδότησης των ΜΜΕ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να προωθήσει τους ευρωπαϊκούς στόχους και να δημιουργήσει τις τεχνικές δυνατότητες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για να επιτρέψει την πρόσβαση των ΜΜΕ στις ε, πηγές αυτές κεφαλαίου. Η κυρία Γκαρντίνη έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, έχει τεράστια σημασία να ενισχυθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο η υποστήριξη στι μικρομεσαίες επιχειρήσει για το ρόλο και τη βαρύτητα που έχουν τον κοινοτικό ιστό σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω υπενθυμήθηκε. Υπενθυμίστηκε ήδη. Και υπενθυμίστηκε ότι είναι οι πραγματικοί πρωταγωνιστέ τη οικονομική ανάκαμψη. Ήθελα να ε, υπογραμμίσω ότι από το 2002 μέχρι το 2008, με τη μεγάλη ανάδειξη του 27 χώρε, δημιούργησαν 9.400.000 νέε θέσει εργασία. Ήδη λοιπόν υπήρξαν οι πραγματικοί κινητήρια δύναμη της απασχόλησης. Τώρα μετά την κρίση έχασαν το 1 τρίτο των θέσεων εργασία που είχαν δημιουργήσει. Και άρα είναι απαραίτητο να σκεφτούμε συγκεκριμένε δομέ, συγκεκριμένα εργαλεία που θα ξαναδώσουν στι μικρομεσαίες επιχειρήσει αυτή την ικανότητα να παράγουν και να δημιουργούν νέε θέσει εργασία. Γιατί αυτό θα έχει όφελο για όλη την κοινωνία. Η πρόσβαση στι πιστώσει ε, είναι ένα από τα σημεία κλειδιά για όλου του επιχειρηματίε. Ε, το 18% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το 2010 ε, απορρίφθηκε ε, η αίτησή τους για δανειοδότηση. Την προηγούμενη χρονιά το ποσοστό αυτό ήταν 12%. Είναι δεδομένα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η πρόσβαση στις ε, ε, πιστοληπτικές ικανότητες ίσως ε, είναι μέρος του Small Business Act που θα περιμένουμε μεγάλη απομονησία να δούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Στην Ιταλία, ε, στο, στην βορειοανατολική περιοχή της Ιταλίας είδαμε μια μεγάλη ανάπτυξη ακριβώς γιατί ένα έξυπνο σύστημα δανειοδότησης υποστήριξε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σας ακολουθήσουμε αυτό το παράδειγμα. Ευχαριστώ. Now I will give the floor to Zoran Thaler for one and a half minute. E, hvala lijepa, gospod predsjednik, gospod komisar Tajani. Rad bi se... Κύριε Σταρέ, ένα μισή λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Tajani? θέλω και εγώ να μιλήσω για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τόνωση της οικονομίας που πρέπει καταρχήν να λαμβάνει υπόψη της τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις διότι δημιουργούν ε, εκατοντάδες εκατομμυρίων θέσεων απασχόλησης Ποια είναι τα βασικά παράπονα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε αυτό το ερώτημα. Πρώτον, είναι η έλλειψη δημοσιονομικής πειθαρχίας. Υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις και δεν λαμβάνουν ε, τα οφειλόμενα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετούμε νέους κανονισμούς σε αυτά τα θέματα και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να γίνουν περισσότερο πειθαρχημένα πλέον, διότι από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Από την κορυφή λοιπόν ξεκινάει το πρόβλημα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θα είχαν προβλήματα αν λάμβαναν τις οφειλόμενες πληρωμές. Επίσης, οι τράπεζες δεν εκπληρούν την αποστολή τους και η ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι όσο υψηλή θα μπορούσε να είναι. τα μέτρα της Επιτροπής, τα οποία μας εξέθεσε και υποστηρίζει και ο κ. Σταγιάννη, θα πρέπει να αποσκοπούν κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει επιτέλους να καλύψουμε τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ευχαριστώ κ. Σκέλη. Ε, ε, ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι καλή βραδιά αυτή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα θέματα που συζητούμε. Ε, έχουν επίπτωση στην πραγματική οικονομία. Συζητήσαμε για τι υπηρεσίε, για τα διπλώματα ευρεσιτεχνία και τώρα για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει, όπω υπόθηκε, έχουν ζωτική σημασία. Ε, από την άποψη της δημιουργίας απασχόληση. Το να δημιουργήσουν θέσει εργασία οι μικρομεσαίε επιχειρήσει δεν είναι δύσκολο, ιδίω αν έχουν πρόσβαση στι πιστώσει. Κάθε εβδομάδα συναντώ επιχειρηματίε, ιδιαίτερα στη χώρα μου, που έχουν πρόβλημα. Ε, το περασμένο Σαββατοκύριακο μια μικρομεσαία επιχείρηση είχε ε, ανάγκη ρευστότητα 4.000 ευρώ και δεν μπορούσε να πάρει ε, το δάνειο. Ε, αυτό το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν αρκεί να επαναλαμβάνουμε ε, το ότι οι τράπεζες είναι πολύ μεγάλες για να χρεοκοπήσουν πρέπει ε, να το αλλάξουμε αυτό το τροπάρι και να το κάνουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντικές για να χρεοκοπήσουν. Αν πάρουν τη σωστή υποστήριξη, κάθε μία από αυτές θα μπορούσε σίγουρα να δημιουργήσει μία επιπλέον θέση εργασίας και με αυτές τις νέες θέσεις εργασίας θα βγούμε από την ύφεση την οποία αντιμετωπίζουμε. Δεν ζητάμε πάρα, πολύ, πάρα πολλά. Συζητώντας τα νέα μέσα για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ε, είναι σίγουρο ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε τα μέτρα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα έχουμε τη διαδικασία Catch the Eye. Η κυρία Μπατζέσκου Ευχαριστώ. Η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα μπορούσε να μας δώσει μία λύση για την οικονομική κρίση. Η ενίσχυση του Small Business Act θα πρέπει να είναι προτεραιότητα και για τα κράτη-μέλη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώνουμε ότι τα τρέχοντα μέτρα δεν έχουν εξαλείψει τα εμπόδια για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Χιλιάδες μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναμένουν θετικά μέτρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης θετικό μέτρο θα ήταν η ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης. Πρέπει να βελτιώσουμε την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά κεφαλαίων για να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για τους επενδυτές. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε την χρηματοδότηση των καινοτόμων εταιριών σε μεγάλη κλίμακα. Η ρουμανική κυβέρνηση πρόκειται να υιοθετήσει ένα πρόγραμμα για την υποβοήθηση της ανάπτυξης μικροεπιχειρήσεων και παροχή κινήτρων σε νέους επιχειρηματίες. Αυτό είναι τμήμα ενός πακέτου κυβερνητικών μέτρων για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ο κύριος Μπατσίτης. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Επίτροπε, η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εξακολουθεί να είναι ένα σημαντικό πρόβλημα παρά τα μέτρα που λαμβάνονται. Είναι κρίσιμη η θέση τους, η κατάστασή τους. Είδαμε την ε, έκθεση του Bankwatch που αναλύει την κατανομή των πιστώσεων της Τράπεζας Επενδύσεων σε τέσσερα κράτη-μέλη και η έκθεση αυτή λέει ότι μέχρι τώρα οι πιστώσεις που δόθηκαν από τις τράπεζες ε, στάθηκαν ε, μόνο για τις ίδιες τις τράπεζες. 50 δισεκατομμύρια ευρώ δόθηκαν για μια διετία και τα κονδύλια αυτά τα έλαβαν οι τράπεζες ε, χωρίς όμως να ενισχυθούν με τα ποσά αυτά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό δείχνει ότι στον τομέα αυτό χρειαζόμαστε πολύ πιο αυστηρό έλεγχο του τραπεζικού τομέα και μεγαλύτερη αρρωγή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα για το θέμα αυτό να πω για αυτά που μα είπε ο Επίτροπος ε, για την χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι σαφέ ότι το κόστο και η διαθεσιμότητα πιστώσεων παραμένει η μοναδική και μεγαλύτερη πρόκληση για τον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη και στην δική μου χώρα, την Ιρλανδία. Πολλέ βιώσιμε εταιρείε συνεχίζουν να έχουν δυσκολίε ε, ε, στο να βρουν χρηματοδότηση από τι τράπεζε, οι οποίε οποία, στην οποία να έχουν ε, πρόσβαση με λογικούς όρους. Ο τομέας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι η ατμομηχανή της ανάπτυξης και της οικονομίας. Ο ιδιωτικός τομέας δημιουργεί τις θέσεις απασχόλησης. Όλα αυτά που κάνουμε εμείς, η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, είναι το να δημιουργούμε το οικονομικό κλίμα που θα οδηγεί σε απασχόληση και σε επενδύσεις και αυτό πρέπει να κάνουμε ε, να δώσουμε ευελιξία και να μην είναι γραφειοκρατική η πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Μετά τη δήλωση του Πρόεδρου της Επιτροπής ε, για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακολουθούμε στενά αυτά τα οποία γίνονται, διότι είπε ο Πρόεδρος ότι θα έχουμε μεγάλη εξοικονόμηση ε, από τις, ε, για την οικονομία και θα πρέπει να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ακριβώς, αυτές που βοηθούν να μειωθεί η ανεργία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γκάλα και κυρία Φιγκορέιντο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κατάσταση των ε, ΜΜΕ σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δραματική, όπου η κρίση τις έχει πλήξει με πολύ σοβαρό τρόπο. Πρέπει να σας πω ότι πολλές ε, δεκάδες, εκατοντάδες μιμιές στην Πορτογαλία έκλεισαν. Πολλές οικογένειες έμειναν στον δρόμο. Αυξήθηκε η φτώχεια, αυξήθηκε η ενεργία. Τα προβλήματα των πιστώσεων των τραπεζιστών, η δυσκολία να έχουν κοινοτικά κονδύλια αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στραγγαλίζει διάφορες επιχειρήσεις και περιοχές ολόκληρες. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει πλήρης μεταστροφή της πολιτικής για αυτές τις περιοχές, ώστε να υποστηριχθούν με αποδοτικό τρόπο αυτές οι ΜΜΕ και να επιμείνουμε με τα δημοσιονομικά συστήματα, ώστε να υπάρχουν προσβάσιμες πιστώσεις και χρηματοδότηση, καθώς και ικανά κονδύλια για αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Ο Κύριε Πρόεδρε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ατμομηχανή της οικονομίας και ο βασικός εργοδότης, γιατί είναι ένας εργοδότης ε, που είναι ο μόνος που μπορεί να δώσει θέσεις απασχόλησης σε περίοδο ύφεση. Εδώ και δεκαετίες έχουμε εμποδίσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης και τους έχουμε δημιουργήσει, τις ε, έχουμε θέσει σε μειονεκτική θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, στην πράξη, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τη Βασιλεία 2 έχουν δυσκολότερη πρόσβαση στο κεφάλαιο. Είναι σημαντική η καινοτομία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να επιβιώσουν. Χρειάζεται όμως χρήματα και έρευνα η καινοτομία. Και γι' αυτό χρειάζεται παροχή κινήτρων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να έχουν καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να επωφεληθούν από τα μέτρα διότι σιγά σιγά εξαντλούνται από την προσπάθεια Ευχαριστώ πολύ και δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Λουάν. Υπάρχουν και στη δική μας χώρα προβλήματα που και στις άλλες χώρες. Πρέπει όμως να πω ότι τα προβλήματα είναι ακόμη χειρότερα σε εμάς. Δεδομένου ότι υπάρχει πρόβλημα πρόσβασης στις πιστώσεις και πρόσβαση σε τεχνικά μέσα και μέτρα που είναι σημαντικά κυρίως όσον αφορά την καινοτομία και την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Θα πρέπει λοιπόν η πρόσβαση στην ενημέρωση ποιότητας να την βελτιώσουμε. Πέρσι το Σεπτέμβριο, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διευκρίνησε ότι το 2011 σχεδιάζεται εμφάνιση στο ίντερνετ των δυνατοτήτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να μπορέσουν να βελτιώσουν τα αποτελέσματά τους. Έτσι θα μπορούν να έχουν δωρεάν παροχή υπηρεσιών, καλύτερη επικοινωνία και καλύτερη γνώση των συστημάτων που υπάρχουν και των χρηματοπιστωτικών δυνατοτήτων. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα του οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα και σε μείωση της γραφειοκρατίας. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εκτίμησα ιδιαίτερα την παρέμβαση του Επιτρόπου κ. Ταγιάννη, γιατί ακριβώς τόνισε το πρωταρχικό πρόβλημα που είναι ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ένα παραγωγικό μοντέλο και άρα ένα κοινωνικό μοντέλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την απασχόληση. Η σημερινή ε, οικονομική κρίση δεν είναι μια παροδική κρίση, είναι μια διαρθρωτική ε, κρίση που βασίζεται, σχετίζεται και με την δομή των αγορών και με την ε, παγκοσμιοποίηση. Η πρόταση ε, του ψηφίσματος θέτει κάποιες προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες, δηλαδή μεγαλύτερη πληροφόρηση όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Πρέπει ε, να γίνουν τα μέσα χρηματοδότησης πιο εύχριστα, τα μέσα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και όπως είπατε, πιο μεγάλη ευελιξία και απλούστευση, ε, μεγαλύτερη, περισσότερη πόρη για την ανάπτυξη και την έρευνα ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να παίξει καθοδητικό ρόλο ε, και οι κανόνες πρέπει να γίνουν πιο σαφείς και κατανοητοί ώστε να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μια, ε, ένα νέο όραμα για τη χρηματοδότηση, διότι την κρίση δεν μπορούν να την πληρώσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά το τραπεζικό σύστημα που δεν κάνει παρά να αυξάνει τα κέρδη του. στο νέο προγραμματισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτές οι απαιτήσει ώστε να αποφύγουμε η ευρωπαϊκή στρατηγική. Διακόπτει ο πρόεδρο, έχετε μόνο ένα λεπτό. Θα πρέπει λοιπόν να περιλαμβάνονται τα απαραίτητα μέσα ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που θέτουμε. Ευχαριστώ. So you had one minute. Συγγνώμη, αλλά είχατε μόνο ένα λεπτό ε, και γι' αυτό σας διάκοψα κύριε Κολίνο. Ήταν η τελευταία μου προειδοποίηση. Ένα λεπτό μόνο έχετε. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Ντανσίλα για ένα λεπτό τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω το γεγονό ότι ακόμη δεν έχουν αρθεί τα εμπόδια για τη βοήθεια των ε, ΜΜΕ στην Ευρώπη. Γι' αυτό θα πρέπει να βελτιωθεί η στρατηγική και να μπορέσουν τα συγκεκριμένα σχέδια και οι δράσεις της Επιτροπής να εφαρμοστούν στα 6 εκατομμύρια μιμιμή που έχουμε, που περιμένουν ε, για να βελτιώσουν τα συστήματά τους, για να βελτιώσουν τα συστήματα καθυστέρησης πληρωμών, για να μειώσουν την γραφειοκρατία. Πρέπει να πω ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πραγματικά μια διέξοδος για την ε, οικονομική κρίση στα πλαίσια της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Θα πρέπει λοιπόν να αποτελέσουν και σε εθνικό και σε κοινωτικό επίπεδο προτεραιότητα. Ευχαριστώ. Έχω άλλον ένα ομιλητή, τον κύριο Σεχέσκη, για, αυτή την, ε, για αυτό το θέμα ή για το επόμενο. Γι' αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι απαιτήσει για μια επιτυχημένη πολιτική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, βρίσκονται στη σωστή λειτουργία τη εσωτερική αγορά. Χρειαζόμαστε σωστή κυκλοφορία όλων χωρίς εμπόδια. Θα πρέπει όλοι να έχουν σωστή πρόσβαση στην αγορά και θα πρέπει οι επιχειρήσεις ε, να είναι έτοιμες για καλύτερο ανταγωνισμό και με μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. θα πρέπει να έχουν ίση μεταχείριση επίσης οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην πρόσβαση στην αγορά. Τα κράτη-μέλη πολλές φορές ε, υποστηρίζονται ορισμένες ε, δικές τους ε, επιχειρήσεις και θα πρέπει να φροντίσουμε την, την ίση μεταχείριση στην Ευρώπη καθώς και τη σταθερότητα των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη. Δεν θα πρέπει παράλληλα να ξεχνάμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό στην ποιότητα ζωής και στο επίπεδο διαβίωσης των απασχολουμένων και των οικογενειών αντιδρούν ίσως λίγο αργότερα στην κρίση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υποστηρίζονται λιγότερο. Αντιθέτως, θα πρέπει να εντείνουμε τη χρηματοδότηση και την υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε κύριε Σικέσκη. Κύριε Επίτροπε, θέλετε να απαντήσετε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η απόψινή συζήτηση τόνισε, όπως φαινόταν και από την πρόταση ψηφίσματος, ότι υπάρχει απόλυτη σύμπνοια ανάμεσα στην βούληση του Κοινοβουλίου και τη βούληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο να ε, τοθεί στο επίκεντρο της ε, οικονομικής πολιτικής για να βγούμε από την κρίση την πραγματική οικονομία και ε, δίνοντας υποστήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι ε, το, το σύστημα των αρτηριών και των φλεβών της οικονομίας μας. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αφοσιωμένη στο να αναζητήσει μια ε, πολιτική λύση στα συγκεκριμένα προβλήματα και χάρη βεβαίως και στην υποστήριξη του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο ε, υιοθετήθηκε η οδηγία για την καθυστέρηση των πληρωμών που είναι πολύ σημαντική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα εμείς πρέπει να πιέσουμε τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν τους ρυθμούς μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Έχουν τέσσερις μήνες από τον Οκτώβριο ξεκινώντας. Θα ευχόμουν όμως τα κράτη-μέλη να ε, ε, επιταχύνουν τη διαδικασία αυτή ε, της ενσωμάτωσης οδηγίας διότι αυτό επηρεάζει και την πρόσβαση στην χρηματοδότηση που στη συνέχεια μπορεί να χρηματοδοτηθεί για την καινοτομία. Μέσω της οδηγίας ε, θα τεθούν σε κυκλοφορία γύρω στα 180 δισεκατομμύρια ευρώ. Ε, δεν πρόκειται όμως μόνο γι' αυτό. Ε, όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις 23 του μηνός θα εγκριθεί η επικαιροποίηση του Small Business Act της Κομισιόν, όπου θα υπάρχουν ε, ε, κάποιες πολύ σημαντικές επιλογές όσον αφορά ε, την ενία θηρίδα για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση που αποτελεί τμήμα των προτάσεων που θα υποβάλουμε στα κράτη-μέλη και επιπλέον θα καλέσουμε όλα τα κράτη-μέλη και όλες τις τοπικές αρχές να διορίσουν τον κύριο ή την κυρία ε, υπεύθυνο, ε, δηλαδή άτομο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στις 16 Φεβρουαρίου θα οριστεί ο νέος υπεύθυνο εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Ντανιέλ Καγιέχα, αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής. Ο κύριος αυτός θα είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της εφαρμογής του Small Business Act και το σημείο αναφοράς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σχετικά με την πολιτική της Κομισιόν. Το κείμενο του Small Business Act θα υιοθετηθεί στις 23 και καλεί ακριβώς όλα τα κράτη-μέλη να κάνουν το ίδιο. Και το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι, μικρομεσ... και οι τοπικές αρχές που έχουν νομοθετική εξουσία. Όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις, η πρόσβαση στις πιστώσεις, μιλήσαμε για το θέμα αυτό, ότι... Ε, ε, ε, ε, ζήτησα λοιπόν ε, ε, να λυθεί το πρόβλημα αυτό διότι προσπαθούμε να βοηθήσουμε να βελτιωθούν οι σχέσεις και ανάμεσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις, ε, ε, στους πιστοτικούς οργανισμούς αλλά και με την, κεντρική, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διότι θα πρέπει να ξεμπλοκάρουμε τα σημεία συμφόρησης ε, και να ξεμπλοκαριστούν τα περίφημα 30 δισεκατομμύρια που έχουν ήδη αποφασιστεί να δοθούν ως δάνεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και που λόγω ε, της δύσκολης μεταφοράς της οδηγίας αυτής στο εθνικό δίκαιο δεν επωφελήθηκαν από το μέτρο αυτό οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, το πρόσφατο Finance Forum ε, ακριβώς τόνισε ε, το πρόβλημα αυτό των σημείων συμφόρησης, δηλαδή που δημιουργούνται ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τις Εθνικές Τράπεζες. Και στην επόμενη συνεδρίαση θα υποβληθεί μια σειρά προτάσεων για το πρόβλημα ακριβώς αυτό. Φυσικά εργαζόμαστε και για το θέμα της απλούστευσης ήδη με συγκεκριμένα μέτρα. Θα σας δώσω ορισμένα παραδείγματα. Ο κανονισμός REACH ζήτησε να μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εφαρμοστικός κανονισμός ε, ενός κανονισμού πάρα πολύ τεχνικού και αυτό είναι ένα μήνυμα που αποστέλουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι έτσι αυτές δεν θα χρειάζεται να προσλάβουν έναν ε, ειδικό ε, μεταφραστή ε, και ειδικό σε θέματα τεχνικά. Γι' αυτό λοιπόν μεταφράζουμε όλη αυτή την νομοθεσία. είναι κάποια τέτοια συγκεκριμένα πράγματα που αφορούν την ε, πλούστευση. Φυσικά θα συνεχίσουν να ισχύουν ε, τα κείμενα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν με το Small Business Act. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την νομοθεσία αυτή και να την εφαρμόζουμε με σοβαρότητα. Και όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και το fitness jack που εισαγάγαμε με την ε, βιομηχανική μας πολιτική και που αφορά επίσης και τα αποτελέσματα που έχει ε, στην ανταγωνιστικότητα η ισχύουσα νομοθεσία ε, και αυτό θα βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν μπορώ παρά να ευχαριστήσω ε, τον κύριο Ρούμπι και να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την έκκληση που μας απευθύνει το Κοινοβούλιο να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση για το επόμενο CHIP 2, CIP 2. δεν μπορώ Τελειώντας, παρανασεγγυηθώ την ε, ε, δέσμευσή μας για όλα αυτά τα πράγματα που είπαμε και να ε, σας πω ότι σε όλες τις ευκαιρίες που μου δόθηκαν ε, ε, διαβεβαιώνω τους πάντες ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι μια προτεραιότητα για μένα. Ούτως ώστε τα γραφειοκρατικά εμπόδια, ε, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, μια πολιτική υποστήριξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να είναι θέματα που θα χαρακτηρίζουν την ε, πολιτική της ε, ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιχειρηματικότητα μέχρι το τέλος της θητείας της. Η υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι για μένα θεμελιώδου σημασίας, διότι όπως είπα και στην αρχή της απάντησής μου, υπάρχει τέλεια σύμπνια απόψεων ανάμεσα σε εσά και εμένα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επιτροπέ. Κλείνει η συζήτηση για το θέμα της χρηματοδότησης των ΜΜΕ και η ψηφοφορία θα γίνει την Τετάρτη το μεσημέρι στις